Um, Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε αν δεν απατώμε πάλι εγκαίρως. Δεν ήρθαν πολλοί, αλλά ευχαριστώ όσους ήρθαν. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν ως πρώτο σημείο την παρουσίαση του κ. Ουφ Γκάινγκοντ, διευθυντή του EMCDDA που θα μας παρουσιάσει δύο εκθέσεις, δύο. Την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ναρκωτικών 2014 και τη Γενική Έκθεση Δραστηριοτήτων 13. Ξέρεις, Wolfgang, ότι υπάρχει και αναμετάδοση για τα νέα δε μέλη. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα των με το οποίο ασχολούμαστε και γι' αυτό παρακαλώ να ενδιαφερθείτε. Uh, λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρη αυτή η παρουσίαση γιατί η Επιτροπή μας η ΕΛΕΦ έχει συναπόφαση για θέματα αντιμετώπισης ναρκωτικών. Οι ψυχοενεργές ουσίες, καινούργιες ψυχοενεργές ουσίες μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα καθώς και ο ορισμός που εμπεριέχεται στην οδηγία για τα ναρκωτικά. Δεν είναι βέβαια εδώ η συγγήτρια, ήταν εχθές, αλλά θα έρθει, θα έρθει μου λένε, θα έρθει σε λίγο. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γκόιτς στην επιτροπή μας. Ορίστε Wolfgang μου και μετά θα ακουστούν ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Για μένα είναι μεγάλη ειδονή η παρουσία μου εδώ απόψε. Ήρθα να σας παρουσιάσω μερικά κύρια σημεία της καινούργια ανάλυσης του EMCDDA για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, η έκθεση για τα ναρκωτικά δημοσιεύτηκε τέλη Μαΐου ήδη αλλά τότε ήταν βέβαια η εκλογική περίοδος για το Κοινοβούλιο και γι' αυτό το λόγο ήρθα τώρα να σας τα πω. Γενικά η ανάλυση μας δείχνει σταθερή κατάσταση με θετικά σημεία σε, μερικά, σε τομείς αλλά και με νέες απειλές για τη δημόσια υγεία και την επιβολή του νόμου και της τάξεως. Ιδιαίτερα βλέπουμε μία τάση μείωσης της χρήσης της ηρωίνης, αλλά τα συνθετικά ναρκωτικά, η κάναβης και τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ναρκωτικά αυξάνονται. Τα σημερινά ναρκωτικά είναι διαφορετικά από εκείνα που γνωρίζαμε μέχρι πριν. Σε γνωστά ναρκωτικά όπως την κάναβη, οι νέες μέθοδοι παραγωγής έχουν αποτελέσματα και για τις ρητίνες και για τα φυτικά προϊόντα. Υπάρχουν πολλές καινούργιες ουσίες λοιπόν. Σημαντική μας ανησυχία είναι ότι υπάρχουν νέα συνθετικά οπιοειδή και παρεστησιογόνα που είναι τόσο δραστήρια ώστε και λίγα μόνο γραμμάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν 10.000 δόσεις. Νέα ψυχοενεργές ουσίες χρησιμοποιούνται και πολλούνται νόμιμα ως σκόνες από την Κίνα και την Ινδία And και εισάγονται στην Ευρώπη και τότε μεταποιούνται και πολλούνται είτε νόμιμα ως ε, προϊόντα έρευνας είτε παράνομα. Παρα, επιτηρούμε πάνω από 400 νέες ψυχοενεργές ουσίες, 81 από αυτές τέσσερις φορές παραπάνω πριν από τέσσερα, από πριν από τέσσερα χρόνια έχουν γίνει γνωστές και αυξάνεται η χρήση τους. Σήμερα ας πούμε 72 ουσίες μας έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα μόνο για αυτό το έτος και που δεν τέλειωσε ακόμα. Επίσης το ίντερνετ παίζει ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση της αγοράς για αυτές τις καινούργιες ψυχοενεργές ουσίες. Το το EMCDDA ταύτισε 650 σελίδες που πουλούν αυτές τις ουσίες στους Ευρωπαίους. Και πέρα από αυτά, νέα πρόκληση για την αστυνομία είναι η πώληση μέσω των λεγόμενων darknet, σκοτεινοδικτύων. Πριν από 15 χρόνια ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν καθώς και χώρες μέλη θέλησαν να δημιουργήσουν ένα νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες ψυχοενεργές ουσίες που τώρα αναγνωρίζεται ως πρότυπο ευέλτης της πρακτικής. Αλλά ο μηχανισμός αυτός τώρα πιέζεται πολύ και λόγω των εξελίξεων που σας ε, περιέγραψα δεν έχει και αρκετούς πόρους ούτε σε κρατικό ούτε σε νοσιακό επίπεδο ούτε στο επίπεδο της οργάνωσής μας. Και φέτος μόνο έξι ουσίες έχουν γίνει αντικείμενο εμβριθούς έρευνας από το EMCDDA και την Επιστημονική του Επιτροπή που αποτελείται από καθηγητάς. Αυτές οι έξι ουσίες λοιπόν φέτος αλλά ε, μελετήθηκαν αλλά μόνο τρεις για την περίοδο 10 με 13. Μόνο τρεις. And the chairman mentioned it already. Όπως σας είπα λοιπόν ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις ψυχοενεργές ουσίες έχει συζητηθεί στην Επιτροπή ΣΕΦ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δεχτεί μία θέση ε, σε δύο έγγραφα. Μία θέση, δύο έγγραφα. Όπως στο παρελθόν, εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε στη διάθεση των δύο εισηγητών και άλλων των άλλων ευρωβουλευτών που θα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Η κάναβης τώρα. Είναι ναρκωτικό όπου πολλώνει την κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει δημόσια συζήτηση που έχει μάλιστα πρόσφατα τροφοδοτηθεί από νομοθετικές αλλαγές σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Λατινική Αμερική. Στην Ευρώπη η κλίμακα της αγοράς της κανάβεως έχει αυξηθεί καθώς και η εγχώρια παραγωγή και είναι γνωστό ότι το ναρκωτικό αυτό χρηματοδοτεί το οργανωμένο έγκολημα. Γενικά η αγορά των παρανόμων ουσιών φαίνεται ότι παραμένει σταθερή. Η κοκαΐνη είναι το κυριότερο τέτοιο ναρκωτικό και οι αμφεταμίνες στις βόρειες και ανατολικές χώρες. Νέες μελέτες για τα πόβλητα και τα ύδατα δείχνουν ότι οι τώρα εμφανίζονται και σε χώρες σαν τη Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρυσι η Ευρωπόλ μας, είπε, μας ανέφερε την ε, καταστροφή στο Βέλγιο των δύο μεγαλύτερων τόπων παραγωγής του έκσταση. Κυρίες και κύριοι, στις ευρωπαϊκές πόλεις το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι πια τόσο ορατό όσο πριν. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις που έκαναν τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Παρόλα αυτά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, παραμένει ακόμα και συνεχώς εξελίσσεται. Μπορώ λοιπόν να σας διασφαλίσω ότι θα συνεχίσουμε να προσέχουμε και να κάνουμε μία έγκαιρη, επίκαιρη και αντικειμενική και ισορροπημένη ανάλυση του προβλήματος των ναρκωτικών. Τώρα, επειδή έχω και δεύτερο θέμα, αυτά είχα να σας πω για την έκθεση για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και έρχομαι τώρα σε μια γενικότερη επιθεώρηση των κυρίων δραστηριοτήτων του EMCDDA το 2013. που εμφανίζονται και στη γενική μας έκθεση πεπραγμένων. Θα μιλήσω λοιπόν για κάποιες από τις βασικές, ε, ε, κάποια από τα βασικά επιτεύγματα και θα σας πω ότι πέρυσι ήταν ένα ειδικό ε, έτος για εμάς γιατί ε, είναι η χρονιά που ε, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο ιδρυτικός κανονισμός μας. Στις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουμε αναπτύξει σημαντικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη ε, για να έχουμε καλή παρακολούθηση των εξελίξεων στο τομέα των ναρκωτικών και φυσικά άμεση απάντηση στις νέες τάσεις και ουσίες. Δημοσιεύσαμε 40 βασικές εκθέσεις αποτελεσμάτων ε, για τους ε, όσους χαράσουν την πολιτική, 34 επιστημονικά άρθρα και Έχουμε και δύο βασικές εκδόσεις, ε, εκδόσεις σταθμό, την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά που σας παρουσίασα και την πρώτη έκθεση για την αγορά των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη στρατηγική ανάλυση που έχει γίνει ποτέ. Όσον αφορά στην έκθεση για τα ναρκωτικά, η πιο σημαντική εξέλιξη το 2013 είναι ότι την ανασυντάξαμε και την εκδώσαμε έξι μήνες νωρίτερα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για το χρονοδιάγραμμα και γιατί θέλαμε οι εκθέσεις ε, να λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες αλλαγές, της τάσεις που γίνονται στον τομέα των ναρκωτικών και τις ανάγκες όπως και τις προσδοκίες του κοινού. Η πλειάδα των πληροφοριών που αναλύουμε και συλλέγουμε τώρα βρίσκεται σε ένα συνολικό πακέτο και βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Μαζί με την Europol λοιπόν εκδώσαμε και την έκθεση για τις αγορές των ναρκωτικών η οποία ε, εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και έγινε σημαντική πηγή αναφοράς για την ανάλυση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με την υπηρεσία μας και τις δικές μας εκδόσεις οι αγορές, η έκθεση για τις αγορές ε, θεωρήθηκε ε, μια πολύ ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό ε, όργανο και έγγραφο και από την ε, Αμερικανική Ένωση των Βιβλιοθηκών. Το 2013 ήμασταν κέντρο πληροφοριών και αριστείας και είχαμε συνδιοργάνωση και οργάνωση πολλών συνεδριάσεων, τεχνικών συναντήσεων πάνω από 25 τέτοιε ε, συνεδριάσεις ειδικών και σχεδόν 280 εκδηλώσεις σχετικά με τα ναρκωτικά έγιναν στην Ευρώπη και αλλού. Έχουμε, δύο, έχουμε πολλά νέα δίκτυα και είμαστε κέντρο αναφοράς για την παροχή πληροφοριών. Ενισχύσαμε τις ε, συνεργασίες μας με άλλους οργανισμούς όπως η Europol. Έχουμε ανταλλαγή μεθοδολογιών και στρατηγικών πληροφοριών και κοινέ στρατηγικές αναλύσεις ε, όπως ας πούμε, την εφαρμογή του EWS. Μαζί με τη CIPOL κάναμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη Eurojust. Πρόσφατα υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για στρατηγικές και τεχνικές πληροφορίες σε τομείς ε, νομοθεσίας και περιοχής ναρκωτικών. Άλλα σημαντικά ε, γραφεία και οργανισμοί είναι το ECDC, το EMA, το FRA Είμαστε πολύ σημαντικοί εταίροι, ειδικότερα στα συστήματα πρόορης ειδοποίησης ε, για τις ψυχοδραστικές ουσίες και υπάρχει και μια ε, νομοθεσία που σχεδιάζεται και την οποία συζητούμε. Επίσης, συνεργαστήκαμε με ιδιωτικού σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Το 2013 συγκεκριμένα συνεργαστήκαμε με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, την Όμιλο Πομπιντού και το ΣΥΚΑΤ που ε, είναι μια συνεργασία των Αμερικανικών πολιτιών και ε, είχαμε συνεργασία με τη Europol και τη Eurostat. Εκτός από αυτή τη ε, συνεργασία, είχαμε και την συνεχή συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες. Και εκτός από αυτή τώρα έχουμε και ένα project με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, τεχνικής βοήθειας, το οποίο έχει σκοπό να τις βοηθήσει να αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης των ναρκωτικών, γιατί αυτό είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013 επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των προκλήσεων, όπως σας είπα πριν, είναι πολύ ε, περισσότερες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων ψυχοδραστικών ουσιών που αν βρήκε το EWS, το σύστημα πρόορης ειδοποίησης, Υπάρχουν σημαντικοί επίσης δείκτες για την παροχή ναρκωτικών που έχουν αναπτυχθεί. Λαμβάνουμε περισσότερα αιτήματα για να λάβουμε μέρος σε σημαντικές ε, συνεδριάσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις δηλαδή. Περισσότερες επίσης επισκέψεις έχουν γίνει στον οργανισμό μας στα κεντρικά γραφεία. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, είχαμε την Επιτροπή Δικαιοσύνης του Δανέζικου Κοινοβουλίου, τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ε, τον ε, Δήμαρχο της Λισαβόνας και τον κύριο Σούλτ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν είναι έκπληξη για σας είμαι σίγουρος ότι να ακούσετε ότι Μέχρι το τέλος του 2013 το 99,74% του οργανισμού μας, ε, του προϋπολογισμού του οργανισμού μας θα έχει ε, δεσμευτεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε τη στρατηγική μας για τα επόμενα τρία έτη, το πρόγραμμα εργασίας 2016-2018. Αυτή τη διαδικασία ε, την έχουμε τροφοδοτήσει με πληροφορίες μέσα από ένα εκτεταμένο ε, δίκτυο διαβουλεύσεων που έχει να κάνει με βασικούς παίχτες στην αγορά και εταίρους όπως ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά το ευρύ κοινό. Ο συνολικός μας στόχος θα είναι να συντελέσουμε σε μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει ενισχύοντας το σύστημα παρακολούθησης, το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται από τα ε, κεντρικά σημεία στα 28 κράτη-μέλη, την Νορβηγία και την Τουρκία και αναλύοντας και περιγράφοντας το φαινόμενο των ναρκωτικών και από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης. Επίσης, θα ε, συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην παρακολούθηση της ε, χρήσης πολυναρκωτικών και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για την παρακολούθηση της κατάχρησης ε, των ε, ναρκωτικών και των φαρμάκων. Θα ενισχύσουμε επίσης τη δυνατότητά μας ε, να έχουμε τεκμηρωμένη δράση μέσα από περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των γρήγορων αντιδράσεων στη χρήση των ναρκωτικών και μέσα από βέλτιστες πρακτικές. Θέλουμε να έχουμε έγκαιρες πληροφορίες, να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης και να επενδύσουμε στην δυνατότητα αξιολόγησης των απειλών που αναφέρεται επίσης και, στην, ε, και στα λίματα και στην ανάλυση Transporter και ένα σύστημα πρόορης ε, προειδοποίησης που ανέφερα πριν. Μετά από τέσσερα χρόνια λοιπόν σταθερής χρήσης του προπολογισμού το 2014 ε, είχαμε μία μείωση 5% σε σχέση με το 2013. Σε αυτά τα πλαίσια ε, ε, και σε μία συνάντηση στη Λισαβόνα, σε μία συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σούλτς μίλησε ε, για την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του οργανισμού μας το 2015. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα είμαι εδώ για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέ, τη εξαιρετική παρουσίαση. Αυτό που είπα στην αρχή, βλέπετε ότι ήρθαν αρκετοί βουλευτές από τότε που ξεκινήσαμε. Είναι μακρύς ο κατάλογος των ομιλητών. Αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρει τους συναδέλφους σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι προφανές ότι εμείς έχουμε έναν εγγενή ρόλο ε, ως κοινοβουλευτική ομάδα για τις νέες ε, ψυχοδραστικές ψυχοτρόπες ουσίες ε, έχουμε να δώσουμε μια γνωμοδότηση ή μάλλον είμαστε στην ε, συνυπεύθυνη και για μια δεύτερη οδηγία θα ακούσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων με βάση τη σειρά που έχουν γράψει στον κατάλογο ξεκινήσουμε τον κύριο Μπόνι μετά η Τερέζα καλό θα ήταν να Είστε στοχευμένοι σε ερωτήσεις σας, γιατί έχουμε μακρό κατάλογο, που είπα. Ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή για την πολύ ξεκαθαρή αυτή παρουσίαση και τις πληροφορίες που μας έδωσε για τις δραστηριότητες ε, παρατηρητηρίου το 2013 αλλά και για το ότι μας περίγραψε και ορισμένες μελλοντικές προκλήσεις. Και τώρα θα μιλήσω πολωνικά. Σας δίνω λίγο χρόνο να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτήν την έκθεση. Βλέπω ότι έχετε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε, δύο θέματα. Μας περιγράψετε δύο νέες στάσεις αλυσίδα ε, προμήθειας ε, ψυχοτρόπων ψυχοδραστικών ουσιών, ρόλος διαδικτύου. Επίσης είναι αρνητικός ο ρόλος του διαδικτύου και έχουμε αυτό το darknet, το σκοτεινό δίκτυο που αναφέρεται. Και επίσης στην έκθεσή σας φαίνεται ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ε, χρήσης συνθετικών οπιοειδών και ψυχοδραστικών ουσιών που είναι εξαιρετικά δραστικές ουσίες. Δηλαδή με απειροελάχιστη ουσία του ναρκωτικού μπορείς να το πολλαπλασιάσεις ε, και να προκύψουν πάρα πολλές δόσεις. Νέο φαινόμενο αυτό και πάρα πολύ δύσκολα ανοιχνεύονται οι έμποροι και το όλο φαινόμενο είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί. Είμαστε περήφανοι στην Ευρώπη όμως γιατί έχουμε σημειώσει επιτυχία σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Το σύστημα που έχουμε λειτουργεί καλά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να τυποποιήσουμε τις πηγές πληροφοριών ώστε να είναι συγκρίσιμα όλα τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στο σύστημα τις διάφορες χώρες. Στην έκθεσή σας λέτε ότι τα δεδομένα των διαφορών χωρών δεν είναι όλα της ίδιας ποιότητας. Ή τέλος πάντων υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και κανόνες για τα παρεχόμενα δεδομένα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης και το κέντρο πρέπει να συνεργαστεί και με υπηρεσίες της Κομισιόν που ασχολούνται είτε με την υγεία είτε με την εσωτερική αγορά. Άρα μπορούν να είναι χρήσιμοι εταίροι σας. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι η έλλειψη διαφάνειας. Πρόκειται για ζούγκλα. Δεν Ξέρει κανείς ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Και από πλευράς κομισιών ε, επιβραδύνεται σημαντικά και η αντίδραση για ανταπόκριση απόκριση των υπηρεσιών της στα αιτήματά σα. Τώρα σε ό,τι αφορά το 2015 ίσως να μην ήταν τόσο βαθιές οι περικοπές Σοφοβόμαστε φοβόμαστε και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως αναφέρατε επίσης πόσες αναλύσεις πρέπει να γίνουν ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς που ελοχεύουν οι κίνδυνοι. Φυσικά και χρειάζονται περισσότεροι πόροι, είναι προφανές αυτό. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συζητούμε τον προπολογισμό του 2016 αυξηθεί αυτός ο προπολογισμό. Έχω οριστεί εισηγητής σε ένα από τα ζητήματα για συναπόφαση για τις νέες αυτές ψυχοδραστικές ουσίες. Ως εισηγητής λοιπόν θέλω να σας πω ότι τον Οκτώβριο νομίζω μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα σας ενημερώσω για τα βήματα που προτιθέμεθα να κάνουμε. Ολοκληρώνω, συνοψίζω. Πρέπει να γίνει τυποποίηση των πηγών πληροφοριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δεύτερο αυτό. Τρίτον, διαφάνεια, ξεκάθαρα να γνωρίζουμε ποιο είναι αρμόδιο γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέταρτον, μεγαλύτερο προπολογισμό. Και πέμπτον, υλοποίηση εφαρμογή όλων των κανόνων σχέση με τα ναρκωτικά. Πρόεδρος Τερέζα, πώς θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα μιλάω ισπανικά. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε και για τα στοιχεία τα οποία μας μετέφερε προφορικά σήμερα το πρωί. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας ε, ευχαριστήσω κύριε Διευθυντά για το έργο που επιτελείτε και εσείς ε, και οι συντροφοί σας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντοπίσει νέες ψυχοτρόπες ουσίες και βέβαια πάνω απ' όλα να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω ότι υπερβολικά συχνά αυτό το κέντρο παρακολούθησης που για μένα είναι ζωτική σημασίας δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σημασία. Δηλαδή, χάνεται μέσα σε αυτό το νηστό, ε, σε αυτό το συνοθήλευμα εκτελεστικών οργανισμών, ε, έχει ένα χαμηλό προφίλ και αυτό το θεωρώ άδικο. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Το είδαμε και όταν ε, έγινε η κατανομή του προπολογισμού των κονδυλίων, είδαμε περικοπές υψηλότερες από άλλους οργανισμούς εγώ δεν το δέχθηκα αυτό, κατέθεσα σχετικά τροπολογίες και ευτυχώς δεν έγινε δεκτή η περικοπή τουλάχιστον στο αρχικό ύψος που προβλεπόταν. Δεν είναι τόσο βαθιές οι περικοπές. Σίγουρα πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερο προεπολισμό Πολύ σωστά είπατε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη δεν έχει επιληθεί. Εξακολουθεί να είναι παρόν. Μπορεί να μην είναι τόσο ορατό γιατί ευτυχώς ε, για τους πολίτες. Ε, υπάρχουν περισσότεροι πόροι και η ίδια η θεραπευτική αντιμετώπιση βελτιώνεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το πρόβλημα. Δεν έχει εξαλειφθεί. Ένα μεγάλο μέρος ε, του προϋπολογισμού έχει ήδη δεσμευτεί σχεδόν όλος ο προϋπολογισμός και είμαστε στην αρχή μόλις. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο τα τελευταία χρόνια οι ψυχοδραστικές ουσίες κερδίζουν έδαφος σε σχέση με πιο παραδοσιακά ναρκωτικά όπως κοκαίνη, ροήνη, Ως εισηγήτρια για την πρόταση οδηγίας με τροποποίηση του, ε, της απόφασης πλαισίου του, 2000, του 2004 για τις ε, ποινές, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τον ορισμό των ναρκωτικών ουσιών, Επεξεργαζόμαστε λοιπόν αυτή την ε, οδηγία. Άλλαξε ο εισηγητής, ο κύριο Μπόνι τώρα είναι αρμόδιο, μίλησε μόλι πριν. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, δεν νομίζω ότι είναι σήμερα το Συμβούλιο παρόν, άρα δεν μπορώ να απευθύνω άμεσα ερωτήσεις στο Συμβούλιο, όμως Ελπίζω ότι καλό θα ήταν ε, να έρθει τουλάχιστον το Συμβούλιο σε μια συνεδρίασή μας και να ακούσουμε τι πρεσβεύει η Ιταλική Προεδρία. Είναι προτεραιότητα για αυτήν αυτό το θέμα. Θέλει να προχωρήσει με αυτές τις διαπραγματεύσεις. Για να δούμε τι γίνεται και με τους τριμερείς διαλόγους και για τον κανονισμό και για την οδηγία. Υποτίθεται ότι έπρεπε να ξεκινήσουν σιγά σιγά. Εγώ πιστεύω ότι, όπως και είπα και πριν, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν από ψυχοτρόπε ψυχοτρόπες ουσίες είναι επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν αν μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση με τα ναρκωτικά αυτά για την επόμενη πενταετία και επόμενη σημαντική ερώτηση, η ταχύτητα και η μεταμόρφωση αυτών των ουσιών και η δικαστική ε, απάντηση, νομική απάντηση να είναι παράνομες αυτές οι ουσίες. Ποιε είναι και ποιε δεν είναι παράνομες όμως γιατί κάποιες δεν είναι από μόνες τους παράνομες, αν αναμειχθούν μεταξύ τους όμως δημιουργείται μια νέωση η οποία είναι παράνομη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη χώρα μου ε, το καλοκαίρι είχαμε κάποιες υποθέσεις με ανθρώπους που δεν ήταν υπήκοοι Ισπανοί, άλλων ε, ε, χωρών υπήκοοι ήταν, αλλά δεν επομένως δεν αφορά το θέμα μόνο εμάς, αλλά και υπηκόους τρίτων χωρών δηλαδή ναρκωτικά που παίρνουν διαφορετικά ονόματα και τέλος πάντων εισήχσε πολύ κοινή γνώμη. Αυτές οι ουσίες ε, μπορούν να δετεθούν πάρα πολύ γρήγορα και κάποιες φορές ε, δεν το γνωρίζουν ούτε τα ε, λεγόμενα βαποράκια ή αυτοί πάντων που τα διανέμουν. Δεν ξέρουν κάποιοι αν είναι παράνομα ή νόμιμα κάποια νόμοι νόμικα ποιοσία που διακινούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς τον Διευθυντή. Πλην της ε, παρακολούθησης και του ελέγχου, τι συστάσεις έχετε να διτυπώσετε προς τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη τι συνιστά αυτό το κέντρο παρακολούθησης ε, σε επίπεδο πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και δι για πολιτικές οι οποίες θα ε, αποτρέψουν ε, τη δράση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν τα ναρκωτικά διασυνοριακά υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος στη δημοσία υγεία από τα διάφορα ναρκωτικά και από αυτές τις νέες ουσίες που αναφέρατε, τα νέα συνθετικά ε, ναρκωτικά, μεθαμφεταμίνες και κάτι ακόμη. Είμαι βέβαιη ότι κάνετε συστάσεις και Τι είδους όμως θέλω να πείτε. Έδρα του κέντρου παρακολουθήσης είναι η Λισαβόνα, είναι στη χώρα μου, είναι η πόλη μου συγκεκριμένα. Τι πιστεύετε, για τις ικανότητες των αρχών ασφαλείας και των αστυνομικών αρχών. Μπορούν πραγματικά να ελέγξουν και να περιορίσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικό σε μια χώρα όπως Πορτογαλία, όπου εδράζεται, όπως ε, σας είπα, το κέντρο παρακολούθησης. Εγώ νομίζω ότι ανεξαρτήτως του τι μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες, οι πόροι, οικονομικοί, τεχνικοί, που έχουν στη διάθεσή τους, κόψαν σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Ενώ στο μεταξύ το οργανωμένο έγκλημα έχει περισσότερους πόρους και μέσα στη διάθεσή του για το λαθρεμπόρο ναρκωτικών. Δεν νομίζω ότι παρακολουθούνται όλα τα αεροδρόμια τόσο καλά στην ε, χώρα μου. Άλλωστε ξέρουμε ότι έγιναν πτήσεις στη CIA και δεν πήρε κανείς μυρωδιά για το τι γίνεται κατά το παρελθόν. Οπότε μπορεί να υπάρχουν αεροπλάνα που προσγειώνονται και να φέρνουν του κόσμου τα ναρκωτικά όλων των ειδών στην Πορτογαλία και κατόπιν στην Ένωση. Ο κύριος Φάιντον Χόζερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την έκθεση, αυτή η δουλειά είναι πολύ σημαντική και δείχνει ε, ότι δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πρόβλημα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν θερμά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την Επιτροπή έχετε πλήρη υποστήριξη όσον αφορά στα οικονομικά μέσα. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η Europol κατάφερε στις 5 ε, Σεπτεμβρίου να βρει ε, και να συλλάβει τόσους ύποπτους. Ήταν πιο μεγάλη επιχείρηση της Europol ε, ε, είναι πάρα πολλά τα άτομα που συνελήφθησαν και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα πρόβλημα όμως που ταυτόχρονα έχει να κάνει και με τη διασυνοριακή διάσταση. Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, καθόλου απλές για αυτό το θέμα. Και όλες οι συζητήσεις που γίνονται πάντοτε αναφέρονται στο θέμα του εμπορίου των αρκονικών από την πλευρά του Ιράν, που είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει κάποια ε, διοχέτευση ουσιών ε, συνεχής και φυσικά οι ιρανικέ αρχές θέλουν την υποστήριξή μας, θέλουν την ε, τεχνική μας βοήθεια. Θέλουμε να τους ε, υποστηρίξουμε λοιπόν για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα αυτά και να ελέγξουν καλύτερα τα ναρκωτικά που περνούν μέσω του Ιράν. Αυτά επίσης ε, τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και με το Αφγανιστάν. Υπάρχει ένα τεράστιο μαζικό εμπόριο ναρκωτικών. Οπότε γενικά ε, θα είναι καλό να έχουμε συνεργασία με τρίτες χώρες, αλλά ειδικότερα με αυτές τις χώρες θα ήταν καλό να έχουμε μια σύσφυξη των ε, σχέσεων και βοήθεια προς χώρες όπως το Ιράν που από μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ, Γιώζεφ. Έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές στον κατάλογο. Ε, το είπα στην αρχή όταν ήταν η αίθουσα άδεια. Απλώς ήθελα να το επαναλάβω ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Το είχα πει στον κύριο και γι' αυτό ακριβώς ε, είναι και τεράστιος ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, κλείνω λοιπόν τον κατάλογο. Να πω ότι ο κύριος ε, Τσούρακ είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ όλοι να τηρείτε τον χρόνο των δύο λεπτών, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της αγοράς των ναρκωτικών. Αυτό που λείπει εδώ παρόλα αυτά είναι μια κοινωνιολογική ανάλυση. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κάτι τέτοιο. Έχετε πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ακούσω κάτι σχετικό. Κάτι που να έχει να κάνει με τις πολιτιστικές αλλαγές ε, που έχουν οδηγήσει στη χρήση των ναρκωτικών και πώς ε, οι κοινωνιολογικές τάσεις συνεισφέρουν στη μείωση της ζήτησης και της χρήσης των ναρκωτικών. Ποιοι είναι οι συσχετισμοί μεταξύ διαφόρων στοιχείων, ε, ας πούμε, πώς είναι η κατάσταση μιας οικογένειας, έχει αυτό σχέση και συσχετίζεται με τη χρήση των ναρκωτικών. Είμαι σίγουρος ότι τέτοια ζητήματα και τέτοιους παράγοντες τους έχετε αναλύσει. Έχετε αναλύσει την αυξητικές και μειωτικές τάσεις στη χρήση των ναρκωτικών. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω επίσης, γιατί εσείς είστε πιο αντικειμενικοί και απαλλαγμένοι από πολιτικές πιέσεις από ό,τι είναι η σε σχέση με την Κομισιόν. Άρα, θεωρείτε ότι θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε κάποια είδη ναρκωτικών. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που τηρήσετε το χρόνο, λέει ο η κυρία Βόζενμπερκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το παρατηρητήριο και τον κύριο Διευθυντή για την λεπτομερή ανάλυση που μας έκανε για αυτό το θέμα. Είμαι νεοεκλεγής αβουλευτής από την Ελλάδα και μάχημη δικηγόρος 32 χρόνια. Έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα των ναρκωτικών και με το θέμα του εγκλήματος στο διαδίκτυο που είχαμε χτες κύριε Πρόεδρε ε, μέρος του οποίου αποτελεί και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Όπως αναφέρθηκε στην έρευνα είδα ότι πραγματικά αναφερθήκατε και στους ιστοτόπους εκείνους που είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί η ταυτότητα είτε του χρήστη είτε του σερβερ διότι πολλές φορές βρίσκονται σε άλλη χώρα από τη χώρα που διαπράτεται το έγκλημα. Έχουν γίνει πραγματικά πολύ σημαντικές πρόοδοι από ό,τι μας ενημερώσατε από το παρατηρητήριο αλλά σίγουρα το πεδίο είναι ανοιχτό ακόμη στην έρευνα για να μπορέσει αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί. Ήθελα να ενημερώσω ότι ένας άλλος τρόπος δυστυχώς διακίνησης, εμπορίου δηλαδή ναρκωτικών γίνεται σε συνδυασμό και με την παράνομη μετανάστευση. Στη χώρα μου όπου η παράνομη μετανάστευση έχει μια έξαρση των μεταναστευτικών ροών, όπω γνωρίζετε, μετά τα γεγονότα στη Συρία και με μετανάστες ε, οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία και είναι πολύ δύσκολη η φύλαξη ιδιαίτερα στα θαλάσσια σύνορα, υπάρχουν εκεί προβλήματα. Εκεί πραγματικά οι ιδιοκτικές αρχέ έχουν συλλάβει διακινητέ ανθρώπων οι οποίοι ταυτόχρονα κάνουν και εμπόριο ναρκωτικών και το κάνουν όχι ω μεμονωμένοι εγκληματίε, αλλά στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματο. δηλαδή μετέχουν σε συμμορίες οι οποίε συστηματικά προβαίνουν σε αυτή τη διακίνηση με τον τρόπο της παράνομης μετανάστευσης. Το βάζω σαν μια παράμετρο που ενδεχομένως να απασχολήσει το παρατηρητήριο. Και τελειώνοντας ήθελα να ρωτήσω ε, κύριε Διευθυντά στα πλαίσια της στρατηγικής που μας αναφερθήκατε για το 2016 18, ε, αν έχετε λάβει υπόψη σας προσωπικά εγώ είμαι πολύ υπέρ της χρηματοδότησης των ενεργειών σας και όλων των ενεργειών που αφορούν σε αυτό το τομέα αλλά το γεγονός ότι σε χώρες του Νότου, όπως τη δική μου χώρα, που βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα λιτότητος και δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν γίνει πολύ σημαντικές περικοπές σε συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή υγείας, ασφάλειας, προστασίας του πολίτη, που είναι συναρμόδια και για την έρευνα και για τη θεραπεία και για την απεξάρτηση και για την πρόληψη στον τομέα των ναρκωτικών και αναφέρομαι σε αυτό διότι αντιλαμβάνεστε ότι η περικοπή κονδυλίων ειδικά στην έρευνα δυσχεραίνει το έργο των αρμοδίων για την αποκάλυψη και νέων ναρκωτικών ούτως ώστε σε επόμενο βήμα να ενταχθούν στην ποινική μεταχείριση αν θα θεωρηθούν ότι σε συνδυασμό με άλλες ναρκωτικές ουσίες αποτελούν και εκείνα ναρκωτικά που απαγορεύονται από τον νόμο ή αν έχουν κάποιες άλλες ιδιότητες και πρέπει να ενταχθούν σε μια άλλη κατηγορία με το δεδομένο όμως ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η διακίνηση ναρκωτικών τελειώνω κύριε Πρόεδρε είναι, χαρακτηρίζεται ως κακούργημα τουλάχιστον αυτό ε, διευκολύνει την διερεύνηση μέσω του διαδικτύου η κακουργηματική μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Uh, next speaker, another colleague Ευχαριστώ. Ένας άλλος συνάδελφος θα πάρει τώρα το λόγο που έχει κάνει και πολλή δουλειά σχέση με τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέιτς. Διάβασα την έκθεσή σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ είμαι στη σοσιαλιστική ομάδα και ασχολούμαι με όλα τα θέματα ναρκωτικών και ψυχοενεργών ουσιών. Και γνωρίζω αρκετά για τις νέες αυτές ουσίες, το οργανωμένο έγκλημα τις διακινεί και φυσικά παράνομα. Στη χώρα μου τη Σουηδία 15 νέοι της περιφέρειάς μου στα νοτιοανατολικά της χώρας την περασμένη εβδομάδα μπήκαν κατεπηγόντως στο νοσοκομείο λόγω της χρήσης ενός νέου ναρκωτικού που λέγεται Σπάιθ και πολύ συχνά η χρήση τέτοιων νέων ουσιών στην αρχή θεωρείται νόμιμη γιατί δεν καταλά έχουμε καταλάβει εγκαίρως πάντοτε ότι είναι παράνομη ουσία. Και αυτό είναι τεράστια απειλή για την νεολαία. Για τους πόρους που διατίθενται απαντήσατε ήδη, είπατε χρειάζονται περισσότεροι. Και στην έκθεση σας επίσης λέτε ότι μερικές χώρες δεν έχουν αρκετά καλό σύστημα εποπτείας ή παρατηρητήρια συστηματικά. Αυτό είναι πρόβλημα διότι πρόκειται για όλο και μεγαλύτερη απειλή προς τη δημόσια υγεία. Για περισσότερη πληροφόρηση λοιπόν από τα κράτη-μέλη μπορούμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία. Ξέρω ότι πολλά προβλήματα αφορούν την ευρωπαϊκή συνεργασία που εξαρτάται, εξαρτάται από την συνεργασία. Ευχαριστούμε η κυρία Στίβενς. Στο πρόεδρε. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, διάβασα στην έκθεση ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πιέζεται πολύ γιατί φέτος ο όγκος στο ύψος των ψυχοενεργών ουσιών έχει αυξηθεί και η διακίνησή του στο εμπόριο επίσης. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής πληροφοριών για τα καινούργια αυτά ναρκωτικά και τις επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όσο έχει τώρα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ή θα έπρεπε να κάνουμε μια αποτίμηση, να το αναθεωρήσουμε, να δούμε μήπως πρέπει να μεταρρυθμισουτεί. Διάβασα λοιπόν την έκθεσή σας και έμαθα ότι υπάρχουν ναρκωτικά που θεωρούνται κουλ cool και σεξι από τους νέους. Το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές είναι παράνομες τις καθιστά ακόμη πιο ελκυστικές για τους νέους. Ίσως λοιπόν να έπρεπε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καμπάνια πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, ειδικά απευθυνόμενη στους νέους. Ίσως πολλές καμπάνιες τέτοιες, όπως είχε γίνει για την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού και υνοπνεύματος. Μήπως θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να κάνουν τίποτα τέτοιο. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Διευθυντή, κυρία Ζολή. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας, πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλά στοιχεία. Θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας την εμπειρία μου και εγώ εργάστηκα στην τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών εδώ και 10 χρόνια από το 81 ζήτησα δεκάδες έτη φυλάκισης για τους ε, λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διαπίστωσα ότι δεν καταλήγουν πουθενά αυτά τα μέτρα. Μετά ασχολήθηκα με το Αφγανιστάν. Ένα συνάδελφος είπε ότι μόλις φύγει το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν θα αυξηθεί εκρηκτικά η παραγωγή οποίου. Η σοδιά του 13 σας το λέω από τώρα, είναι ήδη υψηλότεροι από όσες είχαν ποτέ σημειωθεί στο Αφγανιστάν και αυτό παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, παρά τις εκατοντάδες χιλιάδων δολαρίων που επενδύθηκαν, παρά τα μαθήματα για την καλλιέργεια ζαφοράς αντί για όπιο, παρά τις δεκάδες θανάτων των ασχολούμενων με την καταπολέμηση. Τι άλλο χρειάζεται για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, ότι η καταπολέμηση των ναρκωτικών δεν λειτουργεί, ότι καταναλώνονται τεράστια ποσά για μηδενικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, έτσι μπορούν τα εγκληματικά δίκτυα να διαθέτουν περισσότερους πόρους, χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και τη μαφία. Δεν καταφέρνουμε να σπάσουμε την αλυσίδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, λογικά, θα έπρεπε μετά από 40 χρόνια αποτυχιών να διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός των χρηστών έχει αυξηθεί γεωμετρικά παρά όσα έχουμε κάνει και ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Παραδείγματο χάρη είναι η καταπολέμηση για το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος από τα ναρκωτικά. Δεν καταφέραμε τίποτα ούτε και σε αυτό. Και καλό τους συναδέλφους να τα δουν όλα αυτά και να καταλάβουμε ότι η νόμιμοποίηση ή η διευθέτηση της πώληση των ναρκωτικών είναι η μόνη λύση. Ευχαριστώ. Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις ε, και πραγματικά ίσως χρειάζεται να έχετε πολύ χρόνο για να απαντήσετε σε όλα αυτά, αλλά κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πρόεδρε, πόσο χρόνο θα μου δώσετε. Προσπάθησα να το αποφύγω να σας ε, δώσω συγκεκριμένο χρόνο. Δείξτε την κατάλληλη ευσυνειδησία τέλος πάντων και κάντε ό,τι μπορείτε. Εντάξει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη αυτή της Επιτροπής, να πω ότι με εκπλήσει, με εντυπωσιάζει αυτό που σημαίνει σήμερα εδώ. Έχω έρθει πάρα πολλέ φορές και πραγματικά δεν έχω δει τόσους πολλούς συμβουλευτές παρόντες άλλη φορά να έχουμε τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια φορά είχα έρθει εδώ και ήταν μόνο τρία άτομα μέσα στην αίθουσα. Τους ρώτησα γιατί δεν τους ενδιαφέρει ο οργανισμός μας και μου είπαν ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν δημιουργούμε και πάλι προβλήματα, αλλά η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ωραία λόγια που χρησιμοποίησατε περισσότεροι για τον οργανισμό μας. Έχω 7 λεπτά λοιπόν και γι' αυτό γρήγορα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα. Κύριε Βούνη, να πω ότι δεν βλέπω τόσο μεγάλη έλλειψη διαφάνειας ε, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με αυτούς και ειδικότερα με την ΣΑΝΚΟ και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικέ υποθέσεις. Η δικαιοσύνη ίσως στο μέλλον να είναι λιγότερο σημαντική γιατί από ό,τι φαίνεται στη Νέα Επιτροπή θα υπάρχει μετακύληση των αρμοδιοτήτων στην, Επιτροπή, στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και υπάρχουν και άλλες ε, γενικές διευθύνσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε όπως η Ταξούντ και άλλες. Τώρα για τις πηγές ε, στα κράτη-μέλη αναφερθήκατε πολύ στην ποιότητα των δεδομένων. Κάνουμε γύρω στις 20 συναντήσεις κάθε χρόνο και συζητούμε με τους συναδέλφους από τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένους ε, τομείς, μεθοδολογίες και στάνταρ για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ε, ένα από τα επιτεύγματά μας μαζί με τους εταίρους μας είναι ότι πλέον ε, μιλούμε μια κοινή γλώσσα και έχουμε πετύχει ένα επίπεδο τυποποίησης που είναι πολύ καλό. Ίσως δεν είναι τέλειο, αλλά είναι πολύ πραγματικά καλό. Επίσης, ε, αναφέρατε πολλοί από εσάς ότι το γραφείο μας, ο οργανισμός μας, ε, δεν ε, λαμβάνει την κατάλληλη προσοχή. Συμφωνώ πλήρως, αλλά βλέπετε, υπάρχει μεγάλη βελτίωση σήμερα και υπάρχουν δύο νομικές βάσεις ήδη. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα σας δώσουμε τις συμβουλές. Εμείς δεν είμαστε παρά αυτοί που εφαρμόζουν τη νομική βάση. Εσείς είστε αυτοί που τη θεσπίζετε. Κάτι πολύ σημαντικό ε, είναι αυτό που άκουσα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των εμπόρων και των dealer. Ε, λαμβάνουμε πολλές φορές ε, τηλεφωνήματα από ανθρώπους που έχουν μαγαζιά και μας λένε μας προσέφεραν σήμερα αυτήν την ουσία, ονομάζεται έτσι, αυτό το μόριο και μου είπανε και οι φίλοι μας ότι μας δίνουν μας δίνουν μια έκπτωση 50% επειδή σύντομα μπορεί να απογορευτεί αυτή η ουσία. Όλα αυτά είναι δίκτυα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Τώρα, ε, μιλήσατε για συστάσεις. Δυστυχώς στον κανονισμό μας δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να κάνω συστάσεις, όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, ε, περικοπές ε, στις αστυνομικές υπηρεσίες ε, και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και σε όλες αυτές τις χώρες. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι οι προπολογισμοί στην Πορτογαλία είναι ε, πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες, όμως είναι χώρα διαμετακόμισης για την κοκαίνη η Πορτογαλία. Τώρα υπάρχει ένας μικρός οργανισμός ε, που έχει δημιουργηθεί από 7 κράτη-μέλη, ονομάζεται Κέντρο ε, Ανάλυσης και Επιχειρήσεων, Θαλάσσιων Επιχειρήσεων για τα Ναρκωτικά και ελέγχει την περιοχή του Ατλαντικού είναι οι χώρες αυτές που χρησιμοποιούν την αστυνομία τους και το ναυτικό τους για να μπορέσουν να ελέγξουν την αγορά των ναρκωτικών και αυτό το γραφείο ε, πραγματικά είναι για μας ε, ένα πολύ καλός εταίρος. Βέβαια περισσότερο επιχειρησιακή είναι η λειτουργία του. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, ακόμα και αν απευθύνομαι σε ερωτήσει που έγιναν στα γερμανικά, να πω ότι έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα και μόνο έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με συνολική δράση και παγκόσμια δράση, ειδικότερα για το Ιράν. Σποραδικά έχουμε κάποιες επαφές με εμπειρογνώμονες από το Ιράν, ειδικότερα στον τομέα της υγείας και ξέρουμε ότι έχουν εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικούς ανθρώπους στο Ιράν και στον τομέα της υγείας ε, ε, είναι πολύ καλή η δουλειά που κάνουν. Πριν από κάποια χρόνια η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πάει στο Ιράν για να δουν πώς μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Άρα μπορεί να μην έχουμε κάποια επίσημη συνεργασία με το Ιράν, αλλά σποραδικά έχουμε επαφές. Τώρα, για την εφαρμογή του νόμου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι το Ιράν μας βοηθά να αποφύγουμε τη διαμετακόμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη όμως το να μιλά κανείς με τους πολιτικούς στο Ιράν είναι δύσκολο. Υπάρχει τόση προπαγάνδα στην περιοχή. Είναι δύσκολο να λάβει κανείς ξεκάθαρη πληροφόρηση. Άρα υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν ακόμη. Και επιπλέον να πω ότι με αυτές τις χώρες κάνουμε μόνο όσα έχει συμφωνήσει η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κάτι άλλο ε, που με ρωτήσατε έχει να κάνει με το πολιτιστικό και κοινωνιολογικό κομμάτι. να πω ότι υπάρχουν στοιχεία όπως ε, η οικογένεια, η κουλτούρα της χρήσης, τέτοιοι παράγοντες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα κράτη-μέλη, επειδή είναι δική τους η ευθύνη, πρέπει πραγματικά να προωθήσουν την πρόληψη. Αργότερα κάποιος είπε ότι θα ήταν καλό να έχουμε μεγάλες εκστρατείες για την πρόληψη. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ της μεγάλης δημοσιότητας γιατί υπάρχει λίγη αξιολόγηση και σίγουρα ε, κάποιες από τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει έδειξαν ότι όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικές αυτές οι καμπάνιες αλλά είναι και αντιπαραγωγικές. Απ' την άλλη όμως ε, το να πάει κανείς σε κάποιες μειονότητες, σε κάποιες γειτονιές να πάει στις ομάδες κινδύνου, όποιες και αν είναι αυτές, ε, και να ξεχνάμε καμιά φορά το πολιτικό ορθρό και να το ορθώ και να κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό γιατί προωθούμε την πρόληψη. Και η περιβαλλοντική πρόληψη όπως ονομάζεται είναι πολύ σημαντική, δηλαδή αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον των ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τις οικογένειες, τα σχολεία, τις γειτονιές. Αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Τώρα για την νομιμοποίηση φυσικά δεν μπορώ να πω τίποτα για την νομιμοποίηση αλλά μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούμε το τι γίνεται στον κόσμο, ειδικότερα τη συζήτηση για την κάναβη. Την παρακολουθούμε πολύ στενά και έχουμε και συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή που ασχολείται με τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης μέσω κάποιων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω λοιπόν ότι σε κυβερνητικό επίπεδο, σε κανένα κράτος μέλος αυτή τη στιγμή δεν συζητείται η νομιμοποίηση, ούτε το βλέπω να έρχεται στο προσεχές μέλλον όμως ε, θα δείτε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τι συμβαίνει στην κοινωνία των πολιτών. Εκεί η συζήτηση αυτή θα παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον από ό,τι πλέζει τώρα. Κυρία Βόζεμπεργκ, η παράνομη μετανάστευση και γενικά η μετανάστευση και τα ναρκωτικά είναι θέμα. Και είχα πολλές συζητήσεις με τον διευθυντή της Frontex για το πώς θα μπορούσαμε να δούμε τη σύνδεση μεταξύ του εμπορίου των ναρκωτικών και του εμπορίου ανθρωπίνων όντων, γιατί ε, οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται και αυτοί ως εμπόρευμα, όπως και τα ναρκωτικά. Και οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα δίκτυα θέλουν να βρουν χρήμα όπως και αν έρθει αυτό στα χέρια τους. Όλη αυτή η, κατάσταση στη Μεσόγειο ε, είναι ένα από το παράδειγμα και είναι δύσκολο κανείς να έχει αποδεκτές ε, πληροφορίες για αυτό το θέμα. Για την Ελλάδα τώρα ε, έχουμε πολύ καλή επαφή με τους εταίρους μας εκεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν περικοπές στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα που είναι δραματικές και έχουμε εξαιρετική συνεργασία, έχουμε εξαιρετικούς εταίρους εκεί και ξέρουμε ότι κάνουν ε, πραγματικά πολύ καλή δουλειά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη αλλά να ξέρετε ότι ούτως ή άλλως η υγεία βρίσκεται υποποίηση στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, το Spice που αναφέρατε είναι μία από τις ουσίες που προέρχεται από φυτά. Είναι συνθετικά κανα... Ε, μικρά κομμάτια ε, φυτών, ε, καναβοειδή τα οποία ε, χρησιμοποιούνται. Έχουμε πραγματικά δει πολλές τέτοιες ε, χρήσεις σε συνθετικά ναρκωτικά, έξι την περασμένη εβδομάδα, δύο αυτήν και φτάσαμε και να διαπιστώσουμε πολλούς θανάτους λόγω αυτών των ουσιών. Ε, σύντομα τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να πω ότι παρακολουθούμε τη διαδικασία πολύ στενά όσον αφορά στην θέσπιση νέης, νέας νομοθεσίας. Νομίζω ότι λίγο πολύ απάντησα στην ερώτηση για την ευαισθητοποίηση. Τώρα για το Αφγανιστάν ε, είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε γιατί όπως σας είπα το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και νομίζω ότι ε, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, ε, αλλά και όλες τις χώρες του κόσμου και δυστυχώς ούτε στην Ευρώπη ούτε εκεί λαμβάνεται ε, σοβαρά υπόψη. Το πρόβλημα είναι στο δρόμο, στην πλευρά των καταναλωτών και αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον των πολιτικών δεν είναι μεγάλο για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει ξεχαστεί προς το παρόν. Και αν δούμε το τι συμβαίνει στον κόσμο, πραγματικά ε, είναι κρίμα γιατί πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ε, αυτό το ζήτημα και αν δείτε τι κάνουμε εμείς ε, θα καταλάβετε ότι εμείς προσπαθούμε να σας δώσουμε όσο πιο καλές πληροφορίες γίνεται για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί απαντήσατε σε όλους. Συνάδελφοι, Φαίνεται το ενδιαφέρον εδώ των μελών και των καινούριων. Έχουμε εμείς την νομοθετική οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά υπάρχει φαίνεται και ενδιαφέρον από και από πιο συγκεκριμένες χώρες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου κλίματος. Θα συζητήσω με τους συντονιστές πότε να ξανακαλέσουμε εδώ το EMCDDA γιατί φάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ νέου για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο θέμα Λοιπόν, έχουμε τώρα μια παρουσίαση από την Κομισιόν. Πώς διαδικαστικό, Τιμόθε, τι είναι. Δεν ακούω από εδώ, λέει ο πρόεδρος. Α, τίποτα. Α, καλά, εντάξει, είναι σιωπηρό διαδικαστικό, καινούριο και αυτό. Τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι μια παρουσίαση από την Κομισιόν κατά τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου περί της δημιουργίας του κοινού συστήματος ασύλου για την Ευρώπη το Κοινοβούλιο θέλησε να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. θεωρώντας ότι η χώρα προέλευσής του είναι η αρμόδια για να εξετάσει πιθανή αίτηση για διεθνή του προστασία. Το Συμβούλιο όμως δεν δεχόταν αυτή τη θέση και τελικά το 8-4 παρέμεινε ως είχε στον κανονισμό του Δουβλίνου, αλλά επειδή επεκρέματο και μία δικαστική προσφυγή συμφώνησαν οι συνομοθέτες να τα αποφασίσει τελικά το δικαστήριο και να συμπεριληφθούν οι αποφάσεις του στο άρθρο 8. Έγινε δήλωση και των τριών οργάνων και μετά από την δήλωση και δέσμευση των τριών οργάνων η Κομισιόν πρότεινε για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια του άρθρου 8 με τις δικαστικές αποφάσεις, με την ομολογία. Θα ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μετά τους σκιώδεις και συνεισηγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν στις 26 Ιουνίου ενέκρινε μία πρόταση για την τροποποίηση του 8.4 του κανονισμού του Δουβλίνου για το καθορισμό της ευθύνης των χωρών μελών για την εξέταση αιτήσεων ασυνόδευτων ανηλίκων. Όπως είπατε και εσείς, η πρόταση δίνει συνέχεια στην πρόσκληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στους τελευταίους τριμερείς διαλόγους για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου εφόσον και όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε στις 6 Ιουνίου 2013 και η πρόταση της Κομισιόν απλώς κωδικοποιεί, συμπεριλαμβάνει την ομολογία στο νέο άρθρο 8. Ούτε τίποτα παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Καταρχήν, σύμφωνα με τη χάρτα των θεμελιωδών που την ανέφερε και το δικαστήριο στην λεγόμενη υπόθεση 1α, θεωρήσαμε ότι τα συμφέροντα του ανηλίκου είναι ο κύριος γνώμονας και δεύτερον οι ασυνόδευτοι ανήλικοι επειδή είναι ιδιαίτερα ευπαθής κατηγορία δεν πρέπει να μεταφέρονται χωρίς σκοπό από τη μία χώρα στην άλλη και η εξέταση των αιτήσεών τους να μην καθυστερεί. Τώρα πιο συγκεκριμένα Βάσει της νομολογίας του δικαστηρίου και της απόφασης του, δύο περιπτώσεις υπάρχουν ανηλίκων που δεν έχουν άλλους συγγενείς στην Ένωση. Πρώτον, αν ο ανήλικος έχει υποβάλει διάφορες αιτήσει για προστασία και στη χώρα μέλος όπου βρίσκεται τη στιγμή της αίτηση αυτή η χώρα θα είναι η υπεύθυνη για να εξετάσει την αίτησή του. 84α. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο ανήλικος είναι παρόν στην επικράτεια μιας χώρας μέλους χωρίς όμως να έχει κάνει αίτηση εκεί. Τότε αυτή η χώρα μέλος πρέπει πρώτα να χορηγήσει την ευκαιρία στον ανήλικο να υποβάλει εκεί αίτηση. 8.4β. Και πάλι εδώ δύο υποκατηγορίες περιπτώσεων. Εάν αφού καταθέσει αίτηση ο ανήλικος αποφασίσει να την υποβάλει, τότε θα παραμείνει σε αυτή τη χώρα μέχρι να διεκπαιρεωθεί η αίτηση. Ή άλλη υποπερίπτωση, αν αποφασίσει ο ενήλικος να μην υποβάλει σε αυτή τη χώρα μέλος αίτηση όπου διαμένει, τότε η υπεύθυνη χώρα θα είναι εκείνη όπου έκανε την πιο πρόσφατη του αίτηση. Και αυτό για την καλύτερη δυνατή προστασία του ανηλίκου. 8.4β3. Εκτός από αυτά τα σενάρια ή τις περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις. Έχουμε διατυπώσει και διάφορους κανόνες για να αποφευθεί κατάχρηση του συστήματος, ιδιαίτερα μέσω καλύτερης πληροφόρησης 8.4 γάμα. Καταληκτικά θα ήθελα να ξανατονίσω ότι οι δύο συνομοθέτες κάλεσαν την Κομισιόν στην αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου να καθορίσει η Επιτροπή σαφέστερα τα πράγματα και τις περιπτώσεις και γι' αυτό υπολογίζουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη δυνατή διεκπαιρέωση και ταχύτερη των υποθέσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Φταίω εγώ εντελώς γιατί ήμουν πάρα πολύ χαλαρός έδωσα το λόγο σε όλους τους άφησα να μιλάνε όσο θέλουν ήταν ενδιαφέρον θέμα για τους αδέλφους λοιπόν τώρα έχω καταρτήσει κατάλογο ομιλητών γιατί έχουμε τον εισηγητή και του σκιώδης έχει και η Ιταλική Προεδρία να ε, μας πει τα δικά της παρακαλώ να είστε σύντομοι όλοι κυρία Βίξτρομ εισηγήτρια έχει πρώτο το λόγο Ευχαριστώ. Στην προηγούμενη εντολή μου συγκίτρια για την αναδιάτυπωση του κανονισμού του Δουβλίνου που εγκρίθηκε όπως ακούσαμε τον Ιούνιο του 2013. Πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά για μένα, για πάνω από τέσσερα χρόνια. Και η ομάδα μου πραγματικά ήταν πολύ κοντά με τον άλλο και είχαμε μια φανταστική συνεργασία μεταξύ μας. Ένα άρθρο όμως ε, δεν μπορέσαμε ε, να το διατυπώσουμε όπως θα θέλαμε και συγκεκριμένα το άρθρο 8.4, δηλαδή ποιο κράτος είναι ε, υπεύθυνο για την εξέταση της ασύλου από ένα συνόδευτο ανήλικο, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη και η σύμβαση του Δουπλίνου Έλεγε εκεί που έχει κάνει αίτηση ο ανήλικος. Πρώτο, κράτος πιο πρόσφατο, δεν ξεκαθαριζόταν αυτό. Και τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, το ερμήνευσαν κάνοντας χρήση του παλαιότερου κανονισμού ως προς το ότι θα πρέπει στο πρώτο κράτος μέλο που έφτασαν οι ανήλικοι εκεί να εξεταστεί η αίτησή τους. Δηλαδή, παιδιά στέλνονταν ε, σαν δέματα, σαν βαλίτσες από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτό θέλαμε να τερματιστεί. Διαπραγματεύσει λοιπόν για τον νέο κανονισμό του Δουβλίνου συμφωνούν και όλε οι χώρε ότι οι πρέπει να γίνουν σαφεί. Δεν συμφωνήσαμε όμως πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ήθελα να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να είναι η χώρα στην οποία έχει υποβάλει την πιο πρόσφατη αίτηση ο ανήλικος. Το Συμβούλιο όμως εξακολουθούσε να θέλει να είναι η χώρα όπου είχε υποβάλει την πρώτη του αίτηση ο ανήλικος και αυτό μας οδήγησε σε διέξοδο για αρκετό χρονικό διάστημα και παρά τις προσπάθειές μας δεν καταλήγαμε πουθενά. Εκεί λοιπόν εμείς ως Κοινοβούλιο έπρεπε πλέον να επιδείξουμε δημιουργικότητα και πραγματικά επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη με την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στην ομάδα μας αυτή. Εκείνη λοιπόν τη χρονική στιγμή των διαπραγματεύσεων εκκρεμούσε μια απόφαση του δικαστηρίου ακριβώς για αυτό το θέμα τους συνόδευτους ανηλίκους και ποια χώρα είναι που πρέπει να αποφασίσει. Και αφού δεν μπορέσαμε εμείς να αποφασίσουμε, είπαμε θα αφήσουμε το κείμενο ω έχει, στον παλιό δηλαδή κανονισμό, με την προσθήκη όμω δεδομένου ότι είναι προς το καλύτερο ε, μέγιστο συμφέρον του ανηλίκου. Κάτι άλλο που κάναμε και δεν ήταν και συνηθισμένο, προσθέσαμε μια κοινή δήλωση που στηρίζεται από Συμβούλιο Κοινόβουλιο και Κομισιόν που αναφέρει ότι άπαξ και εκδοθεί απόφαση στο δικαστήριο για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξανανοίξει το άρθρο αυτό στον κανονισμό του Δουβλίνου και να επανέλθει με πρόταση συγκεκριμένη σε εμά που θα λαμβάνει υπόψη τη την απόφαση του δικαστήριου. Με άλλα λόγια, το δικαστήριο αποφάσισε αυτό που εμεί από πολιτική πλευρά δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε. Τον Ιούνιο συγκεκριμένα το 2013, πριν την έγκριση του κανονισμού του Δουβλίνου, αποφάσισε το δικαστήριο. Η απόφαση σημάδιζε απόλυτα με τη θέση Συμβουλίου, μάλλον Κοινοβουλίου και Κομισιόν, θα πρέπει η με τα κινήσεις των αντίκων οι αχρήστες να αποφεύγονται και ότι θα πρέπει το κράτος όπου ο ανήλικος έχει υποβάλει την πιο πρόσφατη αίτηση να είναι αυτό το οποίο θα την επεξεργαστεί. Προτάθηκε λοιπόν ε, νέα ε, εκδοχή τον Ιούνιο από την Κομισιόν και εμείς πρέπει το συντομότερο δυνατόν να την εγκρίνουμε. Χωρίς αμφιβολία πάντοτε πρέπει να δούμε με γνώμονα το των συμφέρον του παιδιού και αυτό το λέει και το 24, το 24 του Χάρτη Μελιδών Δικαιωμάτων. Επίσης, στην απόφαση του δικαστηρίου επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι άκρος ευάλωτα άτομα εξού και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρονται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Χαιρετίζω λοιπόν ε, την πρόταση της Κομισιόν. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή διότι λαμβάνει υπόψη ε, την απόφαση του δικαστηρίου όπως και εμείς συμφωνήσαμε στην κοινή μας δήλωση και ελπίζω να μπορέσει η αλλαγή αυτή του κανονισμού να εγκριθεί τάχιστα. Τρεις σκιώδεις εισηγητές ήταν σκιώδη συζητέ και για τον κανονισμό του Δουβλίνου, η Σιλβί Γκυγιόμ, ο Τίμωθη Κέρκοπ και η Τζιν Λάμπερτ συγκεκριμένα. ξέρουν πολύ καλά λοιπόν περί τίνο πρόκειται και σήμερα είμαι πολύ ικανοποιημένη ε, που δέχομαι τη Ρομπέρτα Μετσόλ, την Μόλι και τη Λάουρα Φερέ, τα τρία νέα μέλη. Και περιμένω να συνεργαστούμε πολύ καλά, να έχουμε μια ομαλή διαδικασία. Ουσιαστικά πρόκειται περί απλής ευθυγράμμισης του κανονισμού με την απόφαση. Δεν θα ξανανοίξουμε κεφάλαια ε, του κανονισμού. Ελπίζω ειλικρινά να έχει την ίδια προσέγγιση προς την πρόταση αυτή και το Συμβούλιο διότι είχαν ήδη δεσμευτεί σε αυτήν την αλλαγή. Και προσβλέπω να συνεργαστώ με την Ιταλική Προεδρία για το θέμα αυτό. Θα επανέλθω σύντομα με την εκθεσή μου προς τους κοιότητες και θα προτείνω και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ Σεσίλια για την συνεισφορά σας και για την ομιλία σας. Θα παρακαλέσω όμως τους υπόλοιπους να είναι πολύ σύντομη γιατί νομίζω ότι η Σεσίλια τα είπε όλα για σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Σεσίλια. Είναι τιμή μου να είμαι ισκιώδης για αυτό το θέμα και να πω από τώρα ότι θα συνεχίσω τη συνεργασία μου όπως ακριβώς έκανε η Άννα Μαρία πριν από μένα. Θα συνεχίσω λοιπόν ε, τη συνεργασία εξ του ΕΛΚ σε αυτό το θέμα. Είναι δύο τα θέματα, όπως είπε η Σεσίλια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των ε, ανηλίκων. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι ανήλικοι που έχουν καταθέσει αιτήσει για άσυλο και πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι ε, αυτά τα παιδιά δεν χρησιμοποιούνται ως πολιτικό μπαλάκι στα κράτη μας. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πολύ αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ, λέω που ήσουν τόσο σύντομη. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Αυτά που είπαμε δείχνουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παραμένουν λεπτό θέμα στις τεταμένες καμιά φορά συζητήσεις που έγιναν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή μεταξύ των δύο οργάνων. Η κοινή δήλωση πάντως υπήρξε και νομίζω καλός και μετά έγινε και η απόφαση, υπάρχει και η απόφαση του δικαστηρίου. Ας μην επανέλθω σε όλα αυτά. Χαίρομαι για την απόφαση του δικαστηρίου και την ερμηνεία που δόθηκε. Τυπικά ήταν τελείως απαραίτητη αυτή η αποσαφήνιση με βάση βέβαια με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του ανηλίκου. Ως προς το περιεχόμενο νομίζω ότι η ευπάθεια της κατηγορίας του ανηλίκου έχει σωστά ληφθεί υπόψη για να αποφεύγονται οι άχρηστες μετακινήσεις. Είναι λοιπόν πολύ καλή η απόφαση. Έχω όμως ένα, μια απορία, μια απορία προς την Κομισιόν. Από την απόφαση και μετά για τις μετακινήσεις των ανηλίκων. Έγινε γνωστό τίποτα νεότερο. Πάντως θέλω να διαβεβαιώσω την κεκυλία για την ε, υποστήριξη από την ομάδα μου. Ευχαριστούμε Σίλβια. Ο σκιώδης των συντηρητικών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορούμε νομίζουμε να πούμε, νομίζω να πούμε ότι και εμείς το υποστηρίζουμε αλλά δεν θέλω να ξεχάσουμε ε, μερικά δευτερεύοντα αλλά ζωτικά θέματα. Ένα από αυτά είναι, συνοδευτικά μάλλον, το πρόβλημα της εκτίμησης της ηλικία, διότι καλό είναι να προστατεύονται οι ανήλικοι και οι νέοι, αλλά έχουμε δει ότι μπορεί να υπάρξει εγκληματική δραστηριότητα που επικαλείται αυτού του είδους την προστασία. Η ηλικία ενός νέου είναι το καθοριστικό στοιχείο εδώ. Πρέπει λοιπόν πρόεδρε, αφού μιλήσαμε για την υποδοχή των νέων που φτάνουν σε μια χώρα και τη μεταχείρισή τους με τρόπο που να μην τους μετακινεί άσκοπα από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά τα πρότυπα υποδοχής νέων στις διάφορες χώρες είναι πολύ διαφορετικά από, τη χώρα, χώρα σε χώρα. Για πολλές χώρες μέλη έχουμε ανησυχίες γιατί φοβάμαι ότι τα πρότυπά τους για τους ανηλίκους ιδιαίτερα δεν είναι αποδεκτά, δεν είναι, είναι απαράδεκτα. Δέχομαι τις γενικές αρχές αλλά νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη όλες θα έχουν το ίδιο υψηλά πρότυπα υποδοχής και δεύτερον να δούμε το θέμα της εκτίμησης της ηλικία. Τέλος, όπως κάθε φορά που αφορά μεταναστευτικά θέματα, θα ήθελα να πω ότι οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι μάλλον για την κακομεταχείριση παιδών, πόσο μάλλον ασυνόδευτων, αυτοί πρέπει να διώκονται από τις αρχές και την Ευρωπόλ και το Frontex ώστε να δικάζονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους δηλαδή για αυτές τις συχνά απαράδεκτες και ανήθικες συμπεριφορές. Δεν πρέπει να υποφέρουν μεν τα παιδιά, αλλά εκείνοι που τους βάζουν σε τέτοια θέση πρέπει να τιμωρούνται. Λοιπόν, η κυρία Μπιόρκ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξει βέβαια αυτό που θα πω. Η ομάδα μας επικρίνει όλο τον κανονισμό του Δουβλίνου. Θα θέλαμε να καταργηθεί τελείως. Αυτή η πρότασή μας συμβαδίζει και με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή την καλύτερη προστασία του ανηλίκου. Και ξέρουμε ότι αυτό στην πράξη δεν γίνεται σεβαστό ούτε από την ομοθεσία ούτε από τις εφαρμαζόμενες διαδικασίες. Ξέρω τι γίνεται στη Σουηδία και νομίζω κάτι ανάλογο συμβαίνει και αλλού, παντού. Χαίρομαι πάντως για την απόφαση του δικαστηρίου και για την πρόταση της Κομισιόν που είναι βελτίωση για τουλάχιστον μία ευπαθή κατηγορία και θα συνεργαστώ και εγώ με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την ε, ταχύτητα. Η Τζιν Λάμπερτ είναι η ισχυώδης για τους πράσινους και είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι πραγματικά με ανακούφισε η κρίση του δικαστηρίου και είναι δύσκολο κανείς να περιμένει μια κρίση για κάτι που σε όλους εμάς εδώ φαίνεται προφανές. Δεν μετακινούμε τα παιδιά πέρα εδώ, θέσα να είναι πακέτα. Συμφωνώ λοιπόν με την εισήγηση ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ε, άμεση διευθέτηση αυτού του ζητήματος, αλλά και με τις ανησυχίες που αναφέρθηκαν από διάφορους συναδέλφους για το πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το θέμα του συμφέροντος του παιδιού και πώς συνεργάζονται τα κράτη-μέλη. Ένα από αυτά τα πράγματα που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς διασφάλισης. Αυτό πολλές φορές είναι πρόβλημα στη μετακίνηση. Η αδυναμία δηλαδή αυτών των μηχανισμών που θέτει σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο τα παιδιά. Υπάρχει κάτι που πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ στενά και ήταν ε, πολύ εύστοχος ο Τίμωθη όταν είπε ότι πραγματικά ε, και η υποδοχή των παιδιών είναι σημαντική γιατί πολλά παιδιά πολλές φορές απάγονται από τις ε, εγκαταστάσεις όπου, φυλάσσονται ή μπορεί να τα κακομεταχειρίζονται. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Ευχαριστούμε την Τίν. Η κυρία Φεράρα, σκιώδες και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη φορά που είμαι σκιώδης και χαίρομαι ε, πολύ που η Σεσίλια και οι άλλοι συνάδελφοι πραγματικά είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούμε. Σίγουρα χρειάζεται να έχουμε ως προτεραιότητα την προστασία του συμφέροντος του παιδιού, των ανηλίκων δηλαδή. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα αποφάσισε το δικαστήριο να γίνονται όσο λιγότερες μετακινήσεις γίνεται και να υπάρχουν και συγκεκριμένα στάνταρ για την υποδοχή που θα εγκρίνουν και θα εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε αυτά τα στάνταρ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τρεις ακόμα ομιλητές. Σας ζητώ να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόταση τη Κομισιόν και στηρίζω και την γραμμή τη εισηγήτρια Σεσίλια Βίξτρομ. Ήμουν ε, εισηγήτρια για το ΕΛΚ, για την έκθεση περί ασυνόδευτων ανηλίκων και είχαμε ζητήσει τότε συγκεκριμένα αυτή η κατάσταση με το πηγενέλα να πάψει. Δημιουργεί μεγάλο στρες και τραύμα στα παιδιά που ήδη είναι ε, με ψυχικά τραύματα λόγω του ότι βρίσκονται συνόδευτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε πει ότι αυτό πηγαίνει αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά κάποιε φορές μάλιστα ε, κρατούνται ε, και δεν ήξεραν ποια είναι η διαδικασία. Ελπίζω λοιπόν να μεταφερθεί η απόφαση αυτού του δικαστηρίου πολύ γρήγορα σε νομοθεσία, να πάψει αυτή η ασάφεια και στη διαδικασία. Το παιδί πρώτα απ' όλα είναι παιδί και μετά μετανάστης. Επίση, ε, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση πληροφόρηση μεταξύ κρατών μελών για το ποιο κράτο είναι υπεύθυνο, αυτό είναι κάτι θετικό. Θα βοηθήσει και στην αποτροπή καταχρήσεων. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να αναφέρω ότι μας ζητήθηκε να συγκροτήσουμε ένα intergroup για τα παιδιά. Ελπίζω να το στηρίξουν ε, οι συνάδελφοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Είναι μια τεράστια τραγωδία, τη βλέπουμε, συμβαίνει στα εξωτερικά μας σύνορα και μόλις ε, φέτος στη Σουηδία δεχθήκαμε 4.000 ανηλίκους ε, ασυνόδευτους από Ιράκ, ε, Συρία. Αυξάνει ο αριθμός συνεχώς. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να στηρίξουν τη συγκρότηση του Intergroup. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Winberg, την επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι πέρυσι η Σουηδία δέχτηκε περίπου 4.000 ασυνόδευτους ανήλικους. Είναι η χώρα με τους περισσότερους. 31% όλων των ασυνόδευτων που φτάνουν στην Ευρώπη έρχονται από τη Σουηδία. Και άρα πολλές φορές χρειάζεται να περάσουν από πέντε άλλες χώρες μέχρι να φτάσουν στη Σουηδία. Αυτό σημαίνει ότι τα άλλα κράτη δεν ενδιαφέρονται αρκετά για την προστασία των παιδών. Πρέπει όλα τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους αντί να αφήνουν τη Γερμανία, την Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία να τα κάνουν όλα. Είναι σημαντικό η απόφαση αυτή για τους ασυνόδευτους ανήλικους να γίνει αντικείμενο κάποιας απόφασης για περισσότερο έλεγχο στα σύνορα του Σέγγεν. Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ολλανδία είναι μια χώρα που έχει δώσει πολλές φορές άσυλο και έχει λάβει και πολλές αιτήσει Παρόλο που ε, τα άτομα συνήθως πρέπει να κάνουν ε, την αίτησή τους ε, στην πρώτη χώρα στην οποία έφτασαν, δεν γίνεται πάντα, έχει να κάνει με τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται. Φυσικά, πολλοί θέλουν να μπουν στην Ολλανδία γιατί είναι πιο εύκολο θεωρούν να μπουν και να κάνουν αίτηση. Οπότε θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Είστε πάντοτε σύντομοι. Μας εκπλήσετε κάθε φορά. Ευχαριστώ. Τέλος, ο κύριος Ντεπλάζη από την Ιταλική Προεδρία. Παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομοι μπορείτε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο και να επιμείνω απλά στο ότι το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Ιταλική Προεδρία. Έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε να εγγυηθούμε την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Όπως σας είπα πρόκειται για ένα θέμα κεφαλαιόδου σημασίας για την Ιταλική Προεδρία. Οι τριμερείς διάλογοι θέλουμε να ξεκινήσουν επί Ιταλικής Προεδρίας. Δεν μπορούμε βέβαια να αναλάβουμε δέσμευση ακόμη γιατί αναμένουμε ακόμη την αντίδραση των κρατών μελών στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά τις επόμενες μέρες θα λάβετε ενημέρωση να βασιστείτε πάντα στην πλήρη συνεργασία μας. Ευχαριστώ το ακολεί πρόεδρο Σεσίλια. Από εσά μια σύντομη ε, δευτερολογία. δέκα δευτερόλεπτα. Χαίρομαι πολύ που έχω αυτού του σκιώδε εισηγητέ στην ομάδα μου και χαίρομαι που και οι σκιώδε εισηγητέ εξέφρασαν τι απόψει των ε, πολιτικών τη ομάδα. Δεύτερον, προ τον Τίμωθη να πω απλά ότι αυτή η αξιολόγηση καλύπτεται στη, στο, στην πρώτη κανονισμό της οδηγίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την νέα τροπολογία, με την ε, αλλαγή του κανονισμού του συγκεκριμένου. Ας το εξετάσουμε ως κάτι τεχνικής φύσεως, μια απλή τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου για να ληφθεί απόψη, υπόψη, συγγνώμη, απόψη του Και πάλι σας ευχαριστώ όλες και όλους. Πρόεδρο Σεσίλια, μπράβο. Έκανε εσύ την, το κλείσιμο ε, ούτε με ρώτησες κιόλας εντάξει μια χαρά τα είπες ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος για να ολοκληρώσω με τη συνάντηση να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις πρώτα απ' όλα 6 Οκτωβρίου την επόμενη εβδομάδα αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε την ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτούς ε, ε, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 6.30 με 9.30 ο Γκίντερ Ρέτιγκερ κοινή ακρόαση με ήτρε Καλ Κλίμπε. Είναι οι επιτρόποι που μας αφορούν. Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 1.30 με 4.30 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που είναι δική μας αποκλειστικά ακρόαση και 1η Οκτωβρίου 9.30 με 4.30 Βυρόβα με Λίμπε και Καλτζούρι Φαμ Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 6.30-9.30 Άντρε Άντσιπ Ίμκο με Λίμπε ως συνδεδεμένη επιτροπή και 3η 7 Οκτωβρίου 9 με 12 το πρωί Φραντ Τίμερμανς Α, όχι, άλλαξε η ώρα. Το απόγευμα θα γίνει η ακρόαση. Θα ήταν κοινή μεταξύ Τζούρι Αύκο Λίμπε η ε, ακρόαση αυτή, αλλά με τη Σοφία που την διακατέχει, η διάσκεψη των πάντων αποφάσισε να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Θα σας ενημερώσουμε, δεν έχουμε ακόμη καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συνεισφορά σας. Γεια σας. Colleagues, a 10 minutes break and then coordinators.